είναι αναπόσπαστο κομμάτι τη ε, Στρατηγική Ευρώπη 2020 που έχουν προσυπογράψει όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ Επίτροπε. Πέρα τη συζήτηση. Θα ψηφίσουμε αύριο στι 12.30. Τώρα, έκθεση Χάντλιτς σχετικά με την ε, διαδικασία μηδέας αξιολόγησης της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Ο εισηγητής έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Σήμερα έχω την τιμή να σας παρουσιάσω αυτή την έκθεση για την διαδικασία της αμοιβαία αξιολόγησης της οδηγίας περί υπηρεσιών. Όπως γνωρίζετε, Επίτροπε, η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ενδιαφέρεται ιδιαίτερα και ζωτικά για το πώς έχουν τα πράγματα για την εφαρμογή, την υλοποίηση της οδηγίας περί υπηρεσιών. Είναι μία από τις οδηγίες, μία από τις πιο σημαντικές νομοθετικές πράξεις πρόσφατα. Γι' αυτό με ιδιαίτερο ενδιαφέρον κοιτάξαμε την διαδικασία αμοιβαία αξιολόγηση και τις προτάσεις για περαιτέρω δράση που στοχεύουν στην ενδυνάμωση, στην ενίσχυση της αγοράς υπηρεσιών στην ΕΕ. Η διαδικασία αμοιβαία αξιολόγηση αφορά τρία σημεία. Πρώτον, την πείρα που αφορά την αμοιβαία αξιολόγηση τη οδηγία περί υπηρεσιών. Δεύτερον, επικεντρώνεται, εστιάζεται στα αποτελέσματα και τι περαιτέρω δράσει που πρέπει να αναλυφθούν για να διευρυνθεί και να εμβαθυνθεί η κοινή υπηρεσία περί υπηρεσιών, η κοινή αγορά υπηρεσιών. Και τρίτον, τι πρέπει να γίνει σε σχέση με μελλοντικά νομοθετικά μέσα και όργανα. Η έκθεση για την αξιολόγηση είναι ένα αξιόλογο μέσο συνεργασίας. Κατέστησε εφικτό στις διοικήσεις των κρατών μελών, στις κρατικές αρχές να μάθουν τι πρέπει να γίνεται για την, τι γίνεται για την εφαρμογή και υλοποίηση αυτής της οδηγίας σε άλλα κράτη και ποιες λύσεις υιοθετούνται. Επίσης σημαίνει πολλές γνώσεις που διαχέονται, που μας δίνουν μια πιο ολοκληρωμένη, παρότι όχι πληρέστατη και απόλυτα ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς μετά από την υλοποίηση, την εφαρμογή της οδηγίας περί υπηρεσιών. Γι' αυτό θεωρούμε ότι χρησιμοποιώντας αυτή τη διαδικασία αμοιβαία αξιολόγησης πρέπει να θεωρήσουμε, να, να πιστέψουμε ότι πρόκειται για κάτι το ευκταίο και επενέσιμο. Ε, επίσης αυτό το μέσο θα πρέπει να χρησιμοποιείται με επιλεκτικό τρόπο και πάντα να εξετάζουμε αναπερίπτωση το τι συμβαίνει σε αναφορά με το, το νομοθετικό έργο. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει η διαφάνεια να διασφαλίζεται και να επαυξάνεται με σε τακτά διαστήματα ενημέρωση των εμπλεκόμενων για το πώς έχουν τα πράγματα. Εμείς σας υποστηρίζουμε την ανάληψη περαιτέρω διαβημάτων και πρωτοβουλειών σε σχέση και με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πάντα με βάση την αμοιβή αξιολόγηση. Επίτροπε, εργαζόμενοι επί αυτής, επ αυτής της έκθεσης ποτέ δεν ξεχάσαμε ότι το πρώτο και κύριο προτεραιότητα στο να δημιουργηθεί μια κοινή αγορά υπηρεσιών είναι μια πλήρης ολοκληρωμένη εφαρμογή της οδηγίας περιπηρεσιών από όλα τα κράτη-μέλη. Και μέχρι σήμερα, δύο χρόνια μετά από αυτή την οδηγία, δυστυχώς δεν έχουμε φτάσει σε αυτή την πλήρη φάση εφαρμογής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελε σε τακτά διαστήματα να ενημερώνεται για το πώς έχουν τα πράγματα όσον αφορά την υλοποίηση, την εφαρμογή αυτών των διατάξεων. Επίσης πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να αναλαμβάνει δράση κατά κρατών μελών που δεν προχωρούν, ώστε να είναι δεσμευτική και υποχρεωτική η εφαρμογή. Αναμένουμε την έκθεση για την οικονομική αξιολόγηση για την, εφαρμο, την υλοποίηση αυτής της οδηγίας. Θα θέλαμε να δούμε αν η εξοικονόμηση που προκύπτει από την εφαρμογή αυτής της οδηγίας πραγματικά επιτυγχάνεται αυτή η εξοικονόμηση και που οι προσδοκίες μας ήταν ίσως υπερβολικές. Όταν αντιμετωπίζουμε οι συζητήσεις για περικοπές και για λιτότητα δεν μπορούμε να χάσουμε τις ευκαιρίες που προσφέρει αυτή η οδηγία. Ιδιαίτερα όταν σε 9 από 10 καινούριε θέσεις απασχόλησης στην ευρωπαϊκή οικονομία βλέπουμε ότι αυτές εντάσσονται στον τομέα των υπηρεσιών. Πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στο να ευθυγραμμίσουμε και να ολοκληρώσουμε την αγορά υπηρεσιών. Εστιαζόμενοι σε τομείς που θα δίνουν τη μεγαλύτερη προστιθέμενη Επίση αξία. Επίσης θα πρέπει πολύ προσεκτικά να δούμε τι τεκταίνεται σε σχέση με την εφαρμογή της ρήτρα για την ελευθερία συναλλαγών. Ίνκο θα ήθελε να εμπλακεί στην διεργασία αυτή εφαρμογής και εποπτείας επιτήρησης της οδηγίας. Θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά ότι έχει τεράστια σημασία. Τεράστια σημασία να διασφαλίζουμε σε αυτή τη χρονική συγκυρία ότι τα σημεία, τα διαμεσα διαμεσολαβητικά θα μπορούν να λειτουργούν σωστά. Single points of operations. Ε, Catch Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πλήρηση, ε, η ε, υλοποίηση της οδηγίας περιπηρεσιών έχει σημαντικό ρόλο για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια σκηνή σε παγκόσμιο πλαίσιο. Ταυτόχρονα μια ολοκληρωμένη υπηρεσία, ε, αγορά για τις υπηρεσίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντική υπόθεση. Οι υπηρεσίες είναι πάνω από δύο τρίτα του ΑΕΠ στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό είναι αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη να ζητήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη να άρουν τα νομοθετικά προσκόμματα και εμπόδια ώστε να μπορεί να λειτουργεί καλά η ενιαία εσωτερική αγορά χωρίς εμπόδια. Στην Ρουμανία γίνονται δοκιμές ε, στον τομέα του τουρισμού και τον οικοδομικό τομέα και άλλους τομείς. Ε, ταυτόχρονα υπάρχει μια ε, υπηρεσία πληροφόρησης, διαμεσολάβησης όσον αφορά την εφικτότητα αυτών στη Ρουμανία. Σα ευχαριστώ και εγώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όπως και η συγγήτρια προηγούμενα ανέφερε, 9 από 10 θέσεις απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της παροχής υπηρεσιών καλύπτονται. Είναι ο κινητήρας της οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με 2 τρίτα συνεισφέρουν στο ΑΕΠ της Ένωσης. Έχουμε την ενιαία εσωτερική αγορά που πρέπει να είναι αποτελεσματική, κύριο μέσο για την οικονομική ανάπτυξη, για τη δημιουργία απασχόληση και διασφάλιση τη ανταγωνιστικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλά απομένουν να γίνουν δυστυχώ ώστε να διασφαλιστεί η καλή λειτουργία αυτού του τομέα και των υπηρεσιών. Γι' αυτό πιστεύω ότι οι τοπικέ αρχέ, περιφερειακέ αρχέ, δημοτικέ αρχέ πρέπει να ενισχυθούν. Πρέπει ο διάλογο με αυτού του θεσμού να αναζητηθεί. Πρέπει να εμβαθύνουμε σε αυτό το διάλογο διάλογο και σε αυτές τις επαφές ε, διότι η διαδικασία της ε, αξιολόγησης, αμοιβαίας αξιολόγησης είναι ένα αξιόλογο μέσο ώστε να ταυτίζονται, να εντοπίζονται προσκόμματα και εμπόδια. Είναι μια κοινή ευθύνη όλων μας και πρέπει να προχωρήσουμε. Εξαρτάται η επίδοσή μας από την εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, βάσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 9 ε, από τις 10 νέες θέσεις εργασίας είναι στον τομέα των υπηρεσιών. Καταλαβαίνετε πόσο κρίσιμη είναι η σημασία του κλάδου για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το παρόν. Διέρχεται μια βαθιά κρίση, ε, γνωρίζει μεγάλη ενεργία η Ευρωπαϊκή Ένωση, επικρατεί ανασφάλεια στην αγορά εργασίας και γι' αυτό το λόγο ε, θα πρέπει τα μέτρα σχετικά με τον τομέα των υπηρεσιών να τηρούνται και να λειτουργούν αισίως ε, σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό προβλέπεται στη ρήτρα αναθεώρηση ε, τη οδηγία ε, περί υπηρεσιών. Η αναθεώρηση αυτή είναι ο μοναδικό μηχανισμός που θα επιτρέψει να λειτουργήσει σωστά η αγορά εργασία ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε. Κυρία Φλασικόβα τώρα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η δημιουργία της ενίας αγοράς για τις υπηρεσίες ε, υπήρξε ένας από τους ακρογωνίους λίθους του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Ε, όμως η αγορά των υπηρεσιών ε, δεν ήταν αυτό τελής αγορά, είχε ως στόχο να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημιουργεί ένα τεράστιο δυναμικό και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτό ως μοχλός για να δημιουργήσει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και για τους εργαζόμενους. Θα πρέπει να δράξουμε αυτή την ευκαιρία κυρίως σε περίοδο κρίσης. Ε, το κράτος όπου παρέχεται η υπηρεσία πολύ συχνά δημιουργεί κολλήματα στους παρόχους υπηρεσιών κυρίως στον ασφαλιστικό τομέα οι ασφάλειες, ε, ε, οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν μπορούν να λειτουργήσουν διασυνοριακά και αντιλαμβάνεστε πόσο προβληματικό είναι αυτό για τις εταιρείες. Ε, θα πρέπει λοιπόν να έρθουν τα συγκεκριμένα προσκόμματα μετά από δράση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να εξασφαλίσουμε μια μεγαλύτερη μάρια για τις επιχειρήσεις και να παρασχεθούν και καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες. Ένωση, σας ευχαριστούμε. Eh. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Ριγογέν. Η δημιουργία μιας αγοράς, ολοκληρωμένης αγοράς ε, υπηρεσιών δεν είναι μόνο η Λίβια, η για την ε, ευρωπαϊκή διαδικασία αποδείχθηκε να είναι ένα απαραίτητο μέλλον για να μπορέσουμε να διευκρινίσουμε αμφίσιμες καταστάσεις που ακόμη υπάρχουν και για να αξιολογήσουμε αν τα μέτρα εγκρίθηκαν από τα κράτη-μέλη και αν εφαρμόστηκαν σύμφωνα με το πνεύμα του νόμου. Επίσης για να μπορέσουμε να επεκτείνουμε τους κανόνες των καλών πρακτικών. Υπάρχουν όμως ακόμη εθνικοί φραγμοί οι οποίοι τροχοπεδούν κυρίως στην ανάπτυξη των επαγγελματικών υπηρεσιών μεταξύ επιχειρήσεων. Πρέπει εμείς να περιφρουρήσουμε ούτως ώστε να εφαρμόζονται σωστά οι διατάξεις της οδηγίας. Η έγκριση της οδηγίας για τις υπηρεσίες αποτέλεσε ορόσημο στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Αλλά η η διαδικασία αμοιβαίας αναγνώρισης μας αποδεικνύει ότι έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας. Ευχαριστώ τελευταίο ομιλητή η κυρία Φιγκερέιδο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εκφράζουμε την θλίψη μας γιατί συνεχίζεται να υπάρχει απελευθέρωση των υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επιδείνωση που υπάρχει σε σχέση με τις οικονομίες των κρατών μελών. Γενικά η ελευθερία ε, εγκατάσταση σημαίνει ότι οι οικονομικές ομάδες και ε, των πιο ανεπτυγμένων κρατών θα εγκατασταθούν με πολύ μεγαλύτερη ευκολία σε χώρες με ευάλωτες οικονομίες και θα συνεισφέρουν για την καταστροφή χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θέσεων απασχόλησης, όπως συμβαίνει στην Πορτογαλία, σε διαφορετικούς τομείς, κυρίως στο εμπόριο, στις υπηρεσίες, και στον τομέα των μεγάλων καταστημάτων και σε άλλους τομείς επίσης. Γι' αυτό ζητούμε, απευθύνουμε έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει τη στρατηγική της για την απελευθέρωση των υπηρεσιών, ώστε να διαφυλαχθεί η απασχόληση, να διαφυλαχθούν οι θέσεις, απασχόληση, οι θέσεις απασχόλησης και η ανάπτυξη των πιο ευάλωτων οικονομιών. Ευχαριστώ. Επίτροπος Άντορ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές. Αυτή η έκθεση για την αμοιβαία αξιολόγηση της οδηγίας για τις υπηρεσίες μας δίνει νέα στοιχεία σχετικά με τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει σε αυτό το τομέα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων της οδηγίας και κατά την περίοδο της μεταφοράς στην Εθνική Νομοθεσία της Οδηγίας. Ε, πιστεύω ότι πρόκειται για μια σημαντική εισφορά στην ε, ποιότητα και σωστή εφαρμογή της οδηγίας σε όλα τα κράτη-μέλη αυτή η έκθεση. Ευχαριστώ την εισηγήτριά μας, την κυρία Μάλγκορζάτα Χάνσλικ, σχετικά με την ανάλυση του ζητήματος και τα ηχηρά μηνύματα που θέλησε να μας περάσει. Ευχαριστώ και τους σκιώδεις εισηγητές, κυρίως την κυρία Εύελιν Κέπχαρτ, ε, που εργάστηκαν με εντυπωσιακό τρόπο για την εφαρμογή της οδηγίας, η οποία εγκρίθηκε το Φεβρουάριο Φεβρουάριο ε, και φυσικά συνεργάστηκαν ε, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την οδηγία, όπως και ο κύριος Χάρμπορ. Ε, καλύπτονται μέσα στην έκθεση όλες οι διαστάσεις της έκθεσης ε, είτε μιλάμε για νομικά ζητήματα ή για πρακτικά ζητήματα και αυτό μας ικανοποιεί. Δεν χρειαζόμαστε μόνο μια προσαρμογή των οικείων νομοθεσιών. Ε, θα πρέπει ταυτόχρονα να μεριμνήσουμε ώστε οι μοναπευθυντικές θηρίδες, τα one-stop shops, τα περίφημα να λειτουργήσουν σωστά και αυτό αναφέρεται με σαφήνεια μέσα στην έκθεση. Επίσης περνάει η συγγήτρια ένα σημαντικό μήνυμα για τα επόμενα βήματα σχετικά με την μια αγορά για τις υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες ε, ε, ε, στο τομέα των υπηρεσιών ήδη υπάρχει μια απτή επιτυχία αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η οικοδόμηση της ενίας αγοράς. Υπάρχει ανεκμετάλλευτο δυναμικό και γι' αυτό θα πρέπει να προχωρήσουμε και η έκθεσή σας συμβάλλει στην επίτευξη αυτού του στόχου. Τον Ιανουάριο του 2011 στην ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει διάφορες προτάσεις για την διαδικασία αμοιβαία αξιολόγηση και τα αποτελέσματα ε, καταδεικνύουν ότι θα πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη τα πρακτικά ε, ζητήματα που θέτουν οι χρήστες, ε, δηλαδή οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Μόνο έτσι θα επιτύχουμε αυτού του στόχου. Ξεκινήσαμε την αναθεώρηση σχετικά με το αν εφαρμόζονται επί που τα νομοθετήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, διαπιστώνεται ότι η πρακτική εφαρμογή τη οδηγία μπορεί επιτόπου να δημιουργήσει προβλήματα. Παραδείγματο χάρη, ένα αρχιτέκτονας που ε, θέλει να εργαστεί στο Βέλγιο μπορεί να υπάγεται στην οδηγία για τι επαγγελματικέ δεξιότητε, στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο και μία σειρά ε, τέτοια ε, από νομικά μέσα που θα πρέπει να εξετάσουμε για να δούμε αν ε, χαρακτηρίζονται από συνοχή. Εξού και κάνουμε αυτήν την ε, δοκιμή, κάνουμε ε, μελέτες στις κατασκευές, στον τουρισμό και στις επιχειρηματικές υπηρεσίες. Σε αυτούς τους τρεις τομείς λοιπόν βρισκόμαστε σε αυτή την πραγματική φάση και τους επόμενους τρεις μήνες μετά τη σύγκριση των αποτελεσμάτων θα επανέλθουμε και το 2012 θα εισηγηθούμε συγκεκριμένες δράσεις ώστε να λειτουργήσει πιο εύρυθμα η ενιαία αγορά των υπηρεσιών. Επιπροσθέτω, ε, θα μελετήσουμε τα ε, συγκεκριμένα ε, προσκόμματα που θα εντοπίσουμε κατά τη διάρκεια αυτή τη αξιολόγηση που σχετίζονται παραδείγματο χάρη με τι απαιτήσει κεφαλική επάρκεια για τι επιχειρήσει. Αυτό σε εθνικό επίπεδο και διασυνοριακά μπορεί να παρεμποδίσει τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης, κυρίω σε τομεί υψηλή προστοθήμενη που όμως μας δημιουργούν ε, πολλές θέσεις απασχόλησης. Ε, δηλαδή φοροτεχνικοί, αρχιτέκτονες, ε, γιατροί, δικηγόροι και ούτω καθεξής. Επίσης παρεμποδίζονται τα καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα χωρίς να ε, εξασφαλίζεται μια επαρκής προστασία για τους καταναλωτές. Θα αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο επιτόπου όλων αυτών των απαιτήσεων ε, που προκύπτουν από το δίκαιο της Ένωσης και το 2012 αν χρειαστεί θα αναλάβουμε νέες πρωτοβουλίες, θα προτείνουμε νέα μέτρα επίσης σε μια μελέτη σχετικά με τις συγκεκριμένες επιπτώσεις οδηγίας ε, για τις υπηρεσίες επί τη βάση των δράσεων που έχουν αναλάβει τα κράτη-μέλη. Μέσα στην έκθεση Αναφέρετε σας αναφέρεται η σημασία που αποδίδει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διεξαγωγή αυτή τη μελέτη και θα ήθελα να σας παρουσιάσω εγώ προσωπικά στις αρχές του 2012 να σας παρουσιάσω τα πορίσματα αυτής της ε, μελέτης. Ε, τώρα, αν ε, εξετάσουμε την αμοιβαία αναγνώριση ως εργαλείο συνεργασίας, ξέρουμε πόσο σημαντικό κομμάτι της οδηγία για τις υπηρεσίες ήταν και ότι συνεπάγεται βαθιές μεταρρυθμίσεις στην οικία νομοθεσία. Αναμφισβήτητα πρόκειται για το εργαλείο του μέλλοντος, όμως ε, συμφωνώ μαζί σας ότι ε, απαιτείται ανάλυση κατά περίπτωση προτού εφαρμόσουμε αυτή τη μεθοδολογία και σε άλλα νομοθετήματα, διότι οφείλουμε να είμαστε ρεαλιστές. Ε, ελπίζουμε να συνεχίσετε να μας υποστηρίξετε για να αξιοποιήσουμε τη δυναμική που έχει δημιουργηθεί από την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πέρα στη συζήτηση θα ψηφίσουμε αύριο στις 12.30.